23 Μαΐου έλεγξε η Επιτροπή η Αρμόδια την εντολή της κυρίας Λίμπερ Βίρινγκ, η οποία ε, από 4 Μαΐου θεωρείται εγκεκριμένη πλέον. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Και άρα λοιπόν...